τρει πράξει, οι οποίε εγκρίθηκαν στα πλαίσια τη ε, συνήθου νομοθετική διαδικασία βάσει του άρθρου 68 του κανονισμού του Κοινοβουλίου. Οι τίτλοι θα δημοσιευθούν στα πρακτικά της ε, παρούσας συνεδρίασης. Να περάσουμε τώρα στην ε,